Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σα συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινή συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Ρωτάτε το σώμα αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού